το 2016-341 ανέφερε λοιπόν αλλαγή η οποία θα πρέπει να εγκριθεί και θα βρείτε το έγγραφο αυτό στα έγγραφα της Ολομέλειας θα δημοσιευθεί το ουσιαστικό έγγραφο με τα έγγραφα, με τα πρακτικά της συνεδρίασης. Δύο γραπτές ε, Διακηρύξεις λάβαμε και υπογράφτησαν από μέρη του Κοινοβουλίου η 7 του 2016 σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της συνεργασίας για τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο και σε ό,τι αφορά την βελτίωση των μηχανισμών ειδοποίησης σε περίπτωση παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο. Ο κύριος Τσεκόφσκι και 18 άλλα μέλη καταφέρουν να συλλέξουν 465 υπογραφές η γραπτή διακήρυξη του κυρίου Καπούτο υπαριθμών 8 2016 για το διαβήτη υπογράφηκε από τον ίδιο και 26 άλλα μέλη και συγκεντρώθηκε 450 υπογραφές και οι διακήρυξεις αυτές θα δημοσιευτούν με τα πρακτικά της συνεδρίασης και θα διαβιβαστούν ε,